στην ημερήσια διάταξη για την κυκλική οικονομία. Ε, δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνω το λόγο και πάλι στον Επίτροπο τον κύριο Τίμερμανς, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Once Σας ευχαριστώ και πάλι. Σήμερα το πρωί εγκρίναμε ένα σημαντικό πακέτο για την ε, κυκλική οικονομία στην Κομισιόν. Είναι από καρπός εντατικής ε, ομαδικής εργασίας και πραγματικά είναι χαρά μου να σας παρουσιάζω αυτό το πακέτο σήμερα εδώ. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο Κατάναν και Έχουμε δουλέψει εδώ και πάνω από ένα χρόνο για να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Γιατί αν θέλουμε αυτή η μετατροπή να γίνει, να, πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς δραστηριότητά μας. Αυτός ο νέο τρόπος εργασίας είναι κάτι που είναι επίσης ο τρόπος για να προχωρήσουμε ε, ως κομισιόν στο μέλλον. Στην εβδομάδα που ξεκίνησε η COP21 στο Παρίσι είναι μια πολύ επίκαιρη ε, ε, πρόταση για την κυκλική οικονομία συνδέεται με τις πολιτικές ενέργειας και κλίματος. Όλα και περισσότερο φαίνονται οι άμεσε επιπτώσει τη κυκλική οικονομία στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν πολύ θετικοί λόγοι να, προφύγουμε, να φύγουμε, να απομακρυνθούμε από το γραμμικό οικονομικό μοντέλο, το οποίο είναι πολύ εντατικό, σε έναν κόσμο που αυξάνεται ο πληθυσμό καθημερινά, όπου ασκείται τεράστια πίεση στη γη, στο νερό, στο τρόφιμα, ε, στα πρώτε ύλε, στην ενέργεια. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να πετάμε μετά. Η κυκλική οικονομία ως θεματολόγια αλλαγή δεν είναι μόνο απαραίτητη για το περιβάλλον, αλλά είναι το μόνο πρότυπο που έχει νόημα μακροπρόθεσμα για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς έχει νόημα να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους με φιέστερο τρόπο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί όσον αφορά τους μισθούς, αν και κάποιες φορές προσπαθεί και το χάνει η Ευρώπη δεν έχει ε, τις ίδιους φυσικούς πόρους όπως άλλα μέρη του κόσμου, γιατί είναι... Ε, είναι ε, πεπερασμένοι οι πόροι μας και εκεί όπου υπάρχουν είναι πολύ ακριβοί. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε ως ε, πρωτοπόρο στην αγορά για τις πράσινες τεχνολογίες. Οπότε δεν είναι το θέμα κατά πόσο θέλουμε να βάλουμε την Ευρώπη σε ένα κυκλικό μονοπάτι ανάπτυξη, αλλά είναι το πώς εμείς στο δικό μας επίπεδο θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες μας και τα κρατημέλη μας να τα καταφέρουν εκεί που θέλουν και χρειάζεται να βρίσκονται, καθώς και να βρεθούν εκεί γρηγορότερα και σε φόρμα Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε συγκεκριμένη όθηση στην κυκλική οικονομία και να επιταχύνουμε τη μετάβαση. Αυτό που παρουσιάζουμε είναι ένα φιλόδοξο και συνολικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό πλαίσιο που πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει δράση και να προχωρήσει προς την ε, κυκλική οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μέσα ε, καινοτομία και κίνητρα. Θα πρέπει να απλοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά σε αυτό το τομέα για να δημιουργήσουμε νέε επιχειρηματικέ ευκαιρίε και να οθήσουμε την αγορά για, τα δευτερεύοντα, ε, για τι δευτερεύουσε πρώτε ύλε. Να είμαστε πιο φιλόδοξοι από το παρελθόν ώστε να ξεπεράσουμε τα απόβλητα με μέτρα που καλύπτουν το σύνολο τη διάρκεια ζωή ενό προϊόντο. Σχεδιασμό, παραγωγή, καλύτερα ενημερωμένη επιλογή κατανάλωση και σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων. Ναι, όλα αυτά με χρηματοπιστωτικά μέσα και ταμεία και κονδύλια. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε με μέτρα αμοιβαία υποστηρικτικά που θα συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο. Θα πρέπει επίση ε, να σας πω δύο λόγια ω ως παράδειγμα για τις προτάσεις μα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ενώ συνεχίζουμε διαρκώ να θέλουμε να προχωρήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων, ε, στην προτεραιότητα αυτή προχωρούμε με την ανακύκλωση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι θα μένουν μέσα στον ίδιο κύκλο και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαρκώ. Τα απόβλητα δεν τα διαχειριζόμαστε όσο καλά θα μπορούσαμε. Από το σύνολο τη παραγωγή των αποβλήτων, μόνο το 36% ανακυκλώθηκε πραγματικά. Το μεγαλύτερο δε μερίδιο, το 37% απλώς στάλει για ταφή ή ε, αποτέφρωση. Μάλλον. Ε, δεν, δεν εκμεταλλευόμαστε το πλήρες δυναμικό ώστε να βελτιωθούν όμως αυτές οι πρακτικές. Χρειάζεται σχετική νομοθεσία. Το νομοθετικό πακέτο που υιοθετήσαμε σήμερα θα προσφέρει ένα, μια, ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής που θα επιτρέψει σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να αναπτύξουν μακροχρόνιες επενδυτικές στρατηγικές που θα εστιάσουν στην πρόληψη, στη νέα χρήση, στην ανακύκλωση ε, και στην αποφυγή της ε, υπερβολικής παραγωγής αποβλήτων και στην την αποτέφρωση είναι φιλόδοξη νομοθεσία και, και μάλλον ε, περιλαμβάνει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ε, για την ε, διαχείριση των αποβλήτων στην εφήλιο. Επίσης θα βελτιωθούν οι, ορισμοί και θα πλουπηθούν οι απαιτήσει αναφοράς. Ψηλές φιλοδοξίες λοιπόν, αλλά λαμβάνουμε υπόψη επίσης τις διάφορες πραγματικότητες καθώς και τις επιδόσεις ανακύκλωσης στην Ένωση. Οι διαφορές σήμερα είναι τεράστιες, ε, αλλά στόχος μας είναι να επιτύχουμε σταδιακή σύγκληση στα επίπεδα καλύτερης πρακτικής. Ε, αυτά θα υποστηριχτούν από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής με 5,5 δις μέχρι το 2020 τα απόβλητα καυσίμων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο μέσο. θέλουμε γρήγορα αλλαγέ, οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά. Είναι απαράδεκτο τόσο πολλά τρόφιμα ε, να σπαταλώνται ετησίως. Στους βιώσιμους ε, αναπτυξιακούς στόχους έχουμε ε, πει ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις απώλειες τροφίμων σε όλες τις αλυσίδες παραγωγής αλλά και προσφοράς και προς αυτό το στόχο θα, θα, αναπτύξουμε αξιόπιστη μέθοδο ώστε να κατανοήσουμε γιατί γίνονται όλες αυτές οι πατάλες και να ε, μειώσουμε τις πατάλες αυτές. Επίσης, ε, ταυτόχρονα θα εργαστούμε μεταξύ των κρατών μελών για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο Κατάινεν. Έχετε το λόγο κύριε Κατάινεν μου κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη η τιμή που συνομιλώ μαζί σας σήμερα για αυτή την σημαντική δέσμη που προτείνει η Κομισιόν. Είναι τμήμα του Ευρω... της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Δέσμης. Η κυκλική οικονομία είναι ένα φαινόμενο που μπορούμε να συγκρίνουμε με την παγκοσμιοποίηση που γνωρίσαμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Δεν είναι απλώς ε, ένα δευτερεύον στοιχείο της οικονομίας είναι ένα, μια τεράστια παγκόσμια τάση και θα συνεχίσει να εμφανίζεται. Οι δέσμοι που προτείναμε είναι πιο φιλόδοξοι από τις προηγούμενες για τα απόβλητα. Τώρα μιλάμε για την ολοκλήρωση του κύκλου, για την πραγματικά κυκλική οικονομία. που είναι θέμα ανταγωνιστικότητας, ανταγωνισμού αλλά και ολοκληρωμένης αγοράς. Αφορά βέβαια εξαρτάται και από την ταχύτητα με την οποία αντιδρούν οι συνομοθέτε. Το θέμα είναι να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να περάσουν από, από μια μη βιώσιμη οικονομία σε μια κυκλική οικονομία αγοράς. Βέβαια η δέσμη αυτή δεν θα μετατρέψει από μια στιγμή στην άλλη από τη γραμμική οικονομία σε κυκλική. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλή αρχή, μια καλή βάση, μια βασική, μια δομή που να προωθήσει την δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας. Τα δύο αρχικά νομοθετήματα για τα απόβλητα θα συμπληρωθούν με αυτό. Υπάρχουν και προτάσεις από το σχεδιασμό των προϊόντων μέχρι το τέλος της ζωής τους. Και θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα τα παράγωγα, τα παράπλευρα προϊόντα. Έτσι θα εμβαθυνθεί η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά που είναι και το σημαντικότερο τμήμα του επενδυτικού μας σχεδίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν φραγμοί που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τη χρησιμοποίηση των πόρων τους και γι' αυτό η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για δευτερεύοντα ε, πρώτες ύλες είναι, είναι σημαντικό θέμα. θέλουμε προϊόντα τα οποία να είναι ας πούμε πιο εύκολο να αλλάξουν και να διορθωθούν αν είναι ελαττωματικά για να υπάρξει μεγαλύτερη έτσι αποτελεσματικότητα. Το eco-design είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να έχουν ισότιμη μεταχείριση καθώς και τις επιχειρήσεις. Η ιδιαίτερη στρατηγική έχει προβλεφθεί για τα πλαστικά Σήμερα μόνο το 25% των πλαστικών αποβλήτων ανακυκλώνονται. Και αυτό έχει πολύ άσχημα περιβαλλοντολογικά αποτελέσματα. Καταλήγει στους ωκεανούς. Θα προσπαθήσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα λύσουμε με βάση τα τελευταία στοιχεία. Επίσης θα αναθεωρηθούν οι κανονισμοί για τα λοιπάσματα. Επίσης, θα υπάρξει νομοθετική πρόταση για τα ελάχιστα πρότυπα για την ε, ανακύκλωση υλικών και για την άρδευση. Αυτά όλα έχουν μεγάλες δυνατότητες για την οικονομία μας και μπορούν να βελτιώσουν το ΑΕΠ μας κατά περίπου, αντιπροσωπεύουν περίπου 20% του ΑΕΠ μας. Θα δημιουργήσουμε επίσης νέα αναθεωρημένα κριτήρια και θα δημιουργήσουμε και παραδείγματα. Τέλος, υποστηρίζουμε την καινοτομία ώστε να υπάρξει η κυκλική οικονομία. Πρέπει να ξανασκεφτούμε τους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης που έχουμε, να δημιουργήσουμε νέα επιχειρησιακά πρότυπα. Στον ορίζοντα 2020 για τη φάση 16 με 20 βάζουμε 650 εκατομμύρια ευρώ για την καινοτομία και 5,5 εκατομμύρια από τα διαρθρωτικά ταμεία για την κυκλική οικονομία. Πέρα από αυτό μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε σχέδια που είναι ή κοινοπραξίε με, με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή καθαρά ιδιωτικά προγράμματα. Γι' αυτό κυρίε και κύριοι, εφαρμόζοντας γρήγορα τις προτάσεις αυτές από τώρα, μπορούμε να πετύχουμε και οικονομικά και περιβαλλοντολογικά ωφέλη αλλά και κοινωνικά τι αυτά. Αλλάζοντας τη γραμμική μας οικονομία σε κύκλικη. Να δώσουμε στους καταναλωτές και καταναλώτριες την ευκαιρία να εφαρμόσουν επιτέλους τις επιλογές τους, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κατάινεν. Και τώρα ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Λαβία από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον αντιπροεδρού που διατήρησαν την υπόσχεση της Κομισιόν και που έθεσαν σε εφαρμογή αυτή την πρόταση που είχαμε εμείς τελήσει το Κοινοβούλιο και την είχαμε περασπιστεί πέρσι. Αυτή η πρόταση την οποία ο αντιπρόεδρος σε την χαρακτήρισε πιο φιλόδοξη, γιατί είναι φιλόδοξη εφόσον πρόκειται για ένα πακέτο για την κυκλική οικονομία και αν θέλαμε να την αξιολογήσουμε μόνο επί τη βάση των στόχων των αποβλήτων θα την αξιολογούσαμε διαφορετικό τρόπο. Αλλά πιστεύω πως είναι πιο φιλόδοξη και γιατί μας δίνει τη δυνατότητα σε θέσεις για τα διαφορετικά κράτη που, έχουν, που ισχύουν διαφορετικές συνθήκες να επιτύχουν στόχους και άρα να έχουν με μια πρόταση πολύ ισορροπημένη σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Ίσως να θέλαμε να ακούσουμε λίγο περισσότερα πράγματα για τα, για τα τρόφιμα απόβλητα. Ε, ακούσαμε κάποια πράγματα, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερα και σίγουρα η διαδικασία θα είναι χρήσιμη για να βελτιωθεί η πρόταση και για να φτάσουμε σε ένα πιο ισορροπημένο πακέτο, όπως το ήθελα και το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Μποναφέ. Η κυρία Μποναφέ, με συγχωρείτε. Κύριε Αντιπρόεδρε, Επίτροπε Εσεί είχατε πει ότι θα παρουσιάσετε τη νέα πρόταση για την κυκλική οικονομία ανάμεσα μέχρι το, πριν το τέλο του χρόνου και σήμερα είστε εδώ και το συζητάμε. Θα προτείνατε μάλιστα μια πρόταση που θα έκλεινε τον κύκλο και δεν θα μιλούσατε μόνο για την ε, ε, ανακύκλωση των ε, αποβλήτων. Σήμερα με συγκεκριμένε προθεσμίε μα προτείνετε συγκεκριμένα βήματα για να επιταχυνθεί η μετάβαση από το οικονομικό μα σύστημα που είναι γραμμικό στο κυκλικό με μια γενική, βασική και θεμελιώδη ε, για εμά τους σοσιαλδημοκράτες. Είναι καλή, καλό σημείο κίνηση. Όμω αυτά τα 600.000 600 τόνοι απόβλητα να μην πετιούνται στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Θα ήταν λάθο να σκεφτούμε ότι η κυκλική οικονομία για την ε, περιβαλλοντική πολιτική ότι είναι μόνο ένα θέμα που αφορά τα απόβλητα. Είναι πολύ περισσότερα. Διάφορε γενικέ διευθύνσει έχουν εργαστεί πάνω σε αυτή την πρόταση και αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι πρόκειται για μια πολιτική mainstream σε όλου του τομεί τη Επιτροπή. Και εμεί θα επιμείνουμε για να υπάρξουν και ε, τα κατάλληλα κονδύλια. Υπάρχει όμω και κάτι ε, το οποίο δεν τηρήσατε απόλυτα την υπόσχεσή σας να μειώσετε το 75% τα αστικά απόβλητα ε, είναι σημαντικό αλλά όχι αρκετό να είναι σαφές. Δεν είμαστε εμείς ε, φανατικοί των στόχων, ε, ούτε ένα, μια ποσοστία μονάδα πάνω ή κάτω. Με ένα δικό χάρτη όμως φιλόδοξο, όπως εσείς παρουσιάσατε, για να είστε αξιόπιστος, θα πρέπει να στηρίζεστε με, ε, να βασίζεστε σε στόχου, οι οποίοι να είναι μετρήσιμοι και να είναι και οι ίδιοι φιλόδοξοι. Και αν θέλουμε πραγματικά κυκλική οικονομία, θα πρέπει να είμαστε το ίδιο φιλόδοξοι, να προτείνουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και αξιόπιστο και θα στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων. Ε, και γι' αυτά όλα δεν θέλουμε εμεί να χαμηλώσουμε το πύχη των προσδοκιών μα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Δεμέσμακερ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρας ή τα απόβλητα είναι πόρος. Εσείς τα είπατε αυτό κύριε Τίμερμανς, πετυχημένο. Ε, καλύτερη και περισσότερη αηφόρος χρήση των πόρων είναι βασική. Έχουμε 1,5 χρόνο καθυστέρηση θα μελετήσω σε λεπτομέρειες την πρότασή σας, αλλά ε, θέλω να ρωτήσω κάτι για την νομοθεσία, για τα απόβλητα. Πρώτον, το είπατε κι εσείς, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών στην υλοποίηση της κείμενης νομοθεσίας και με τους στόχους 2020. Στη Φλάνδρα ανακυκλώνουμε εμείς 65% των αστικών και οικιακών αποβλήτων, ενώ κάποια άλλα κράτη-μέλη ρίχνουν στις χωματερές ακόμα το 80%. Τι θα γίνει με αυτή τη ε, διαφορά, αυτό το χάσμα ε, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, κλείσει. Δεύτερον, ξέρω ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο, αλλά έχουν μειωθεί οι φιλοδοξίες μας από το, για το 2030 από 70% στο 65%. Αυτό είναι πρόκληση για πολλά κράτη-μέλη και δεν είναι τόσο καλή επιλογή. Υπάρχουν άλλες λύσεις για να συμφωνήσουν όλοι. Για παράδειγμα, ε, ενδιάμεση στόχη, προγράμματα αδελφοποίησης κτλ. Τρίτον, ε, κανόνες δεν χρειάζονται μόνο για χώρες που δυσκολεύονται, αλλά και για πρωτοπόρους, όπως είναι η δική μου περιφέρεια. Πώς θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει καινοτομία εδώ. Και τέλος, η απαγόρευση υγειονομικής ε, ταφής ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει επιγόντως να έρθει. Πώς θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. τώρα... Ε, και τηρήσατε και το χρόνο σας. Ο κύριος Γκεμπράντι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο υπήρξε μια πολιτική γκάφα Αποσύρθηκε το πακέτο για τα απόβλητα και τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Μια νέα νομοθετική πρόταση που είναι πιο αδύναμη από την προηγούμενη και υποθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένει από το Κοινοβούλιο να αυξήσει το επίπεδο και να κάνει αυτή τη μάχη με το Συμβούλιο. Εγώ είμαι πρόθυμος κύριε Επίτροπε να το κάνω, αλλά έχουμε και ένα πρόγραμμα δράσης. Δράσεις. Πού είναι οι δράσεις. Μόνο στο κτίριο Μπερλεμόν περιορίζεται αυτό στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ε, μία αντιγραφή και μάλιστα αποδυναμωμένη της πρότασης του 2011. Άρα δεν έχουμε δύο χρόνια, αλλά τέσσερα καθυστέρηση. Μετά από όλα αυτά τα στεναρά και τα βαρύγδουπα που ακούσαμε από τους επιτρόπους, να ε, επιταχύνουμε για την κυκλική οικονομία φοβούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει με το παρόν πρόγραμμα δράσης. Ε, ε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόνω να επιταχύνει και ουσιαστικά, όχι μόνο στα λόγια. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Χουαρίς Διαμπάουνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμανς, κύριε Κατάινεν, η πρότασή σας ε, αφίσταται από εκείνη του Κοινοβουλίου, απομακρύνεται. Δεν υπάρχει ε, συγκεκριμένη πρόταση για μέτρα και για ελοποίηση και αυτό φρενάρει ε, τη δυνατότητα που έχουμε για συστηματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια γνήσια κυκλική οικονομία που μεταξύ άλλων θα εξαφανίσει τελείως τα τελικά απόβλητα. Οποιαδήποτε επένδυση εκεί θα πρέπει να ε, ανταποκρίνεται στην ανακύκλωση. Δηλαδή να μην υπάρχει πουθενά επένδυση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ε, σκουπιδιών που να μην αιτιολογείται. Δηλαδή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και μόνο. Εγώ σας ζητώ περισσότερη φιλοδοξία στην πρόληψη και στην επαναχρησιμοποίηση. Τα βιολογικά απόβλητα να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται. Αυτό είναι απολύτως εφικτό και ε, υποφελές παντού. Και μπορούν η Λουμπιάνα, η Γκουιπούσκουα, η Κονταρίνα ε, που το έχουν ήδη πράξει να σας βάλουν τα γυαλιά. Ευχαριστώ. Ε, λέει η Πρόεδρος, το λόγο έχει ο κύριος Κλέρτς. Για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Τίμερμανς. Εκπληρώσατε την υπόσχεσή σας ότι μέχρι τα τέλη του 2015 θα έχουμε τη δέσμη για την κυκλική οικονομία. Την έχουμε τώρα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι πιο φιλόδοξο από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες δέσμες. Χάσαμε πολύ χρόνο ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι θα εφαρμοστεί πράγματι σαν δρόμος του μέλλοντος η κυκλική οικονομία. Υπάρχουν βέβαια και θετικά σημεία, αλλά και ελλείψεις, ελλείψεις. Η αποδοτικότητα, καλύτερη χρήση των πόρων και οι δείκτες που επέβαλε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η μείωση της μόλυνσης στη θάλασσα και η μείωση της πατάλησης των τροφίμων σας υπενθυμίζω ότι τον Ιούλιο φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ψήφισε όλα αυτά, αλλά χάθηκαν φαίνεται οι προτάσεις αυτές στους διαδρόμους της Κομισιόν. Δεν ακούσαμε τίποτα πολύ καινούριο. Είναι μία επαναδιατύπωση της οδηγίας για τα απόβλητα. Και όλα τα υπόλοιπα είναι μέτρα μη συγκεκριμένα, ασαφή. Κύριε Τίμερμανς, ποια εγγύηση δίνει η Κομισιόν ώστε η δέσμη αυτή πραγματικά να εφαρμοστεί. Ποια είναι αυτή η αγορά την οποία αναφέρεται που θα είναι λέει εγγύηση της εφαρμογής αφού δεν υπάρχει ακόμα τέτοια αγορά. Λέτε ότι τα απόβλητα θα ανακυκλώνονται και θα γίνουν ενέργεια. Αυτό είναι κάτι που μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δεν χρειαζόμαστε την αποτέφρωση. Έτσι υπαστρέφουμε στην εποχή, στην παλαιολιθική εποχή, ίσως και στην νεολιθική. Κάνατε ορισμένες καλές προτάσεις, επιτρέψατε χώρες που μπορούν να εκπληρώσουν αυτούς τους στόχους, αλλά πώς θα το πράξουν όταν πούν, όταν δηλώσουν ότι δεν μπορούν να τους εκπληρώσουν. Ότι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους. Ε, Monsieur Pellicini, s'il vous plaît, pour euh, une minute au nom de l'EFDD. Grazie, Presidente. Ah, κύριος Πελιτσίνη, Καμία αναφορά στην εξάλληψη των κινήτρων για τα ορυκτά καύσιμα. Κανένα στόχος για την ε, νέα, για την ε, νέα χρήση. Κανένα στόχος όσον αφορά ε, τους ε, συσκευασίες που περνά από το 80% στο 75%. Ένα στόχος για τα απόβλητα τροφίμα από το 35% πάει στη καμία υποχρέωση. Εγώ από τότε που είμαι εδώ αυτό που άκουσα περισσότερο είναι η λέξη φιλοδοξία. Είναι αυτή η λέξη όμως που έχει χάσει το περισσότερο της νόημα όσον με αφορά. Γι' αυτό οι βουλευτές που γίνονται συνένοχοι και που χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη για να περιγράψουν την έκθεσή σας, την πρότασή σας, είναι συνένοχοι σε μια αποδυναμωμένη πρόταση. Ένα λεπτό, ο κύριος Λίζε τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταθέτει σήμερα την πρόταση. Αυτό είναι το αποφασιστικό. Είναι πιο φιλόδοξη, ερωτηματικό. Εν πάση περιπτώσει είναι διαφορετική η πρόταση. Θα πρέπει να την αναλύσουμε και συμφωνώ με όλους εκείνους που μιλούν για τις πατάλη τροφίμων που ήθελαν και περίμεναν λίγα περισσότερα και θα έρθουν οι σχετικές τροπολογίες να μην αμφιβάλλεται. Χρειάζεται δουλειά σε αυτή την πρόταση για πολλούς λόγους. Να πω κάτι επίκαιρο για την προστασία του κλίματος. Εάν καταλήγει στη χωματερή ε, το σκουπίδι, βγαίνει μεθάνιο, το οποίο μεθάνιο είναι χειρότερο αέριο του θερμοκηπίου από το διοξίδιο του άνθρακα. Γι' αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε. Στη Γερμανία 20% ένας ολόκληρος κλάδος της οικονομίας προέρχεται από την ε, ανακύκλωση. Ε, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα μελετήσουμε την πρόταση, αλλά πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά και να μην κάνουμε απλώς συζητήσεις αρχής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Παρνιό, για ένα λεπτό. Εγώ το έχω γράψει αυτό στην έκθεσή μου για την COP21. Αυτή η COP21 και η Σύνοδος Κορυφής των Παρισίων δεν έχει στόχο μόνο να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά να αλλάξουμε υπόδειγμα στην οικονομία. Η κυκλική οικονομία λοιπόν θα βοηθήσει να αλλάξουμε μυαλά και ε, είναι ενδιαφέρον ε, να δούμε αυτή την πρόταση οδηγίας που βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αντιλέγω. Για να κάνουμε οικονομίες στις πρώτες ύλες, 630 ε, δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εμπορικό έλλειμμα ε, οφείλεται στην εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Και για το περιβάλλον 48% το 2030 και 83% το 2050 θα πέσουν σε σύγκριση με το 12 εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ιδού λοιπόν τα ωφέλη της κυκλικής οικονομίας, καλές οι προτάσεις και σύμφωνες με το δικό μας στόχο που αυτή τη στιγμή συζητείται στο Παρίσι στην COP21. Ο κύριος Χένκελ, για ένα λεπτό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στη συζήτηση αυτή γιατί ήμουν και πρώην μάνατζερ του ΒΒΕΦ στη Γερμανία και πρώην πρόεδρος του ΣΕΦ της Γερμανίας των βιομηχάνων, είναι ότι πολύ συχνά εδώ προβάλλουμε ιδεολογικά επιχειρήματα και ασχολούμαστε με αυτά, αντί να ασχολούμαστε με τα επιστημονικά επιχειρήματα. Αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης πλαστικού, PVC, που ορισμένοι εδώ στο Κοινοβούλιο θέλουν οπωσδήποτε να το καίνε. Μα είναι δυνατόν αυτό αντιτίθεται στην ίδια την ιδέα της κυκλικής οικονομίας. Μέχρι το έτος 2030 σε μια κυκλική οικονομία μπορούμε να εξοικονομήσουμε 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα έρχεται το Σέτερομ σένζιο το ευρώ, θα πρέπει να καταργηθεί γιατί οδηγεί σε διχόνοια στην Ευρώπη και σε διαπληκτισμούς. Ο κύριος Σεβίσκα, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε και Επίτροπη, ας κοιτάξουμε τι λέει το παρόν κείμενο και η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διχαστεί, η νομοθεσία έχει φρακάρει στο Συμβούλιο, έχουμε κράτη-μέλη με πολύ κακές επιδόσεις στη διαχείριση των αποβλήτων έχουμε ε, πλαστογράφηση δεδομένων, δεν έχουμε ενιαίους ορισμούς και πάει λέγοντας. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι μια συνολική θεώρηση. Μια συνολική, το υπογραμμίζω και χαίρομαι γι' αυτό. Μπορούμε να συζητήσουμε τους αριθμούς 65% και τα λοιπά, αλλά θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, ε, να ε, έχουμε μια αντίληψη, ένα σχεδιασμό, ένα κόνσεπτ και να το εφαρμόσουμε. Και δεν νομίζω ότι ε, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που σας επικρίνουν. Δύο σχόλια να κάνω. Πρώτον, οι ορισμοί και οι στατιστικές και τα στοιχεία δεν θα είναι εύκολο. Αλλά πέρα από τα οικονομικά κίνητρα που δίδονται, πέντε δεύτερα, ας κοιτάξουμε λίγο και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για φορολογικά και άλλα κίνητρα, γιατί αυτό είναι ευρύτερο. Συγγνώμη, πρέπει να τελειώσω. Ελπίζω στο μέλλον να έχω περισσότερο χρόνο, γιατί έχω και άλλες ιδέες να πω. Ευχαριστώ κύριε Φλόρεντς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ δεν είμαι δυσαρεστημένος, ήμουν πολύ δυσαρεστημένος όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε την έκθεση, τηρήσατε το λόγο σας και τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες. Ωραία. Τώρα έχει καταλάβει και ο πολίτης και η πολιτική ότι είναι σημαντικός ε, κλάδος, ο κλάδος των φυσικών πόρων. Μεγάλο ρόλο παίζουν εδώ οι μέρες και τα ποσοστά ακούω. Παρακαλώ να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Γιατί αν δεν έχουμε μέθοδο και κριτήριο πώς θα φτάσουμε στους στόχους δεν έχουν νόημα οι αριθμοί. Στη, στην ε, Γερμανία μπορεί να εμφανίζονται πολύ καλές επιδόσεις και στην Ιταλία κακές, αλλά ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης μπορεί να ισχύει το αντίστροφο. Ας ε, ασχοληθούμε λοιπόν με την ανακύκλωση, με την κυκλική οικονομία. Για το πρόγραμμα δράσης θα ήθελα λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Και εκεί, κύριε Αντιπρόεδρε, θα πρέπει να εργαστείτε σκληρά για να υπάρξει ένα συνολικό πακέτο, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Κύριος Παολούτσι, για ένα λεπτό. Grazie, signora Presidente. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, το πακέτο και η ανακοίνωση για την κυκλική οικονομία αποτελούν βήμα μπροστά. Μας αρέσει η προσέγγιση του συστήματος που ξεπερνά μια λανθασμένη προσέγγιση ε, της ε, εξοικονόμησης και πρόκειται για πράσινους διαγωνισμούς, για διαχείριση βιώσιμη των αποβλήτων. Όλα αυτά είναι καλά. Βέβαια στην ουσία μας ικανοποιούν πολλά αλλά δεν είναι και όλα εντάξει. Θα πρέπει οι στόχοι να επιτευχθούν γρήγορα, γιατί ο χρόνο είναι σημαντικό. Χρειάζεται περισσότερο θάρρο και αποφασιστικότητα, δηλαδή το αντίθετο από αυτό που έκανε το Συμβούλιο στην υπόθεση Volkswagen. Πιο φιλόδοξοι στόχοι για τα απόβλητα, πιο δεσμευτικοί χρόνοι και προθεσμίε για του στόχου. δείκτε αποτελεσματικότητα και επιδόσεων, ε, δέσμευση να στηριχθεί η απόφαση τη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για μείωση στο μισό το των, ε, της πατάλης τροφίμων, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την επιτεύξη αυτών των στόχων. Ο κ. Ζιμπ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν σήμερα ενέκρινε ένα σύνολο φιλόδοξων μέτρων. Οι στόχοι που ορίστηκαν ειδικά όσον αφορά την ανακύκλωση είναι καλή, είναι μια πρόοδος σε σχέση με τις προηγούμενες διατάξεις, ωστόσο θα πρέπει να το τονίσουμε ότι αυτό το σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συμφωνία και συνεργασία με τις τοπικές με συγχωρείτε αρχές και την κοινωνία γιατί ε, αυτοί οι στόχοι λέγαμε ότι δεν θα εξασφαλίσουν τόση απασχόληση όσο το προηγούμενο πρόγραμμα, όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει επίσης να ε, λάβουμε υπόψη ένα σημαντικό σημείο, ότι δηλαδή την ανακύκλωση των τοξικών προϊόντων. Κάποιος ανέφερε το πλαστικό. Σήμερα πολλά πλαστικά πηγαίνουν στα σκουπίδια, πάνε προς τα φύ. Αλλά πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να δώσουμε σε, αυτές τις, σε κάποιες χώρες ίσως πέντε χρόνια παραπάνω, αλλά να επιτύχουν τους στόχους 100%. Ε, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το τελευταίο καιρό οι διάφορες διαδοχικές συγκρούσεις και οι παγκόσμιες κρίσεις δεν, μπόρεσαν να, δεν μας άφησαν να, να καλλιεργήσουμε ελπίδες και εμπιστοσύνη στο μέλλον. Ε, ακόμα ένας λόγος για να υπογραμμίσουμε την ε, σημασία της πολιτικής συνένεσης ε, ενώπιον αυτής της διάσκεψης για το κλίμα στο Παρίσι. Το μήνυμα του Παρισιού είναι παρόμοιο με το μήνυμα αυτού του πακέτου της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι και οι πλανήτες θα πρέπει να μπουν στο κέντρο της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι θα μπορέσουμε να λύσουμε θέματα κλειδιά όπως η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόληση, η μείωση των ισοτήτων, η διατήρηση των ε, ωκεανών και η προστασία της βιοποικιλότητας. Ε, μπορούμε να έχουμε ελπίδα και να είμαστε αισιοδοξοί. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την γραφειοκρατία και τα λάθη εφαρμογή να ε, επηρεάσουν τόσο σημαντικές στρατηγικές και αποφασιστικές. Η θα πρέπει οι πολίτες να υιοθετήσουν αυτή την, πρόοδο, αυτή την πορεία ως δική τους και να ε, επιτύχουμε έτσι πρόοδο. Ευχαριστώ. Κύριο Σταγιάννη, σας ευχαριστώ Επίτροπε, εκπρόσωποι της Επιτροπής για να εγγυηθούμε βιώσιμη ανάπτυξη στην Ένωση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά με πιο ευφύ τρόπο. Η κυκλική οικονομία αντιπροσωπεύει μια ανάγκη για την Ευρώπη. Πρέπει να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξίδιου του άνθρακα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ακόμα και στον τομέα της, των εφοδιασμού πρώτων υλών. Η κυκλική οικονομία είναι μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Θα βοηθήσει τι επιχειρήσει μα να είναι πιο ανταγωνιστικές, θα ανοίξουν αγορές, θα υπάρξει ανάπτυξη και σε παραδοσιακούς τομείς όπως ο χάλιβας και το αλουμίνιο και θα δοθούν κίνητρα στην πράσινη οικονομία. Θετικά δέχομαι λοιπόν το πακέτο της Κομισιόν που στόχο έχει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο κινητοποιώντα την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων Αυτό το πακέτο λοιπόν αποτελεί ένα ακόμα βήμα τη στρατηγική επαναβιομηχανοποίηση τη Ένωση, που ενέκρινε η Κομισιόν με στόχο το 20% ε, ακατέργαστου εγχώριου προϊόντος ε, από το βιομηχανικό τομέα. Δεν μπορούμε παρά να θυμόμαστε το κεντρικό ρόλο της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Σε ευχαριστώ. Έχετε μπλε κάρτα κύριε Ταγιάννη, τη δέχεστε. Από τον κύριο Σάνι. Κύριε, Γιάννη, ε, κύριε Ταγιάννη, συγγνώμη, δέχεστε ε, τη μπλε κάρτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ταγιάννη, αναφερθήκατε σε δύο σημαντικά θέματα για το πρασίνισμα της βιομηχανίας και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πώς αυτά δαπανώνται. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κυκλική οικονομία έχει περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλέον εκτήματα. Ας πούμε, ε, τα χρησιμοποιημένα και φθαρμένα ελαστικά αυτοκινήτων. Συχνά με ευρωπαϊκή ενίσχυση ε, αυτά χρησιμοποιούνται περισσότερο και μολύνουν, ρηπαίνουν ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Ε, βέβαια θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Αυτό προσπαθούσα πάντοτε να πετύχω όσο ήμουν επίτροπος. Η ισορροπία ανάμεσα στη βιομηχανική και στην περιβαλλοντική πολιτική. Μπορεί να είναι είναι σίγουρο ότι θα είναι επιτυχία κάτι τέτοιο. Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση δεν μπορεί παρά να είναι πράσινη. Πρέπει φυσικά να βρούμε ανά τομέα τις σωστές για να ευνοήσουμε τη βιομηχανία χωρίς να βλάπτουμε το περιβάλλον. Κάτσε δι' Μάλετιτς, κυρία Μάλετιτς πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε πρώτε αντιπρόεδρε. Συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να γίνει ανταγωνισμός μεταξύ μισθωτών αλλά με, για την καλύτερη χρήση των πόρων. Με τους πόρους που διαθέτουμε να γίνει καλύτερη χρήση και καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων ή των ουσιών που μέχρι τώρα αποβάλαμε. Η πρόταση είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και δείχνει ότι στην πρώτη θέση βάζουμε την καλή διαχείριση των πόρων μας και των προϊόντων μας. Ο στόχος Zero Waste είναι πολύ σημαντικός, αλλά χωρίς να χρησιμοποιείται η αποτέφρωση. Τέλος, τα 6 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε με το οικολογικό design, το eco-design, είναι επίσης κάτι το οποίο βρίσκουμε πολύ θετικό. Κύριος Καπούτο, η νέα πρόταση της Κομισιόν για την κυκλική οικονομία σέβεται τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ενώπιον του Κοινοβουλίου. Το πακέτο είναι λίγο λιγότερο φιλόδοξο και υπάρχουν και κάποιες ε, ε, κάποιες απώλειες, ας πούμε, κάποιες ε, πράγματα που ξεχάστηκαν. Ε, στην Κομισιόν παραμένουμε στο 65% μείωση των αποβλήτων. Ενώ είχαμε πει για μείωση ε, κάθε είδους διάλυσης και κάθε είδους ταφής οι οικονομικές και καταναλωτικές συνήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αβίωτο πρότυπο όσον αφορά το περιβάλλον. Εμείς ζούμε σε πιο ευημερή περιοχή του κόσμου και γι' αυτό έχουμε την ηθική υποχρέωση να αναπτύσσουμε προϊόντα και διαδικασίες ε, κομμένες και ραμμένες ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την κυκλική οικονομία και να προχωρήσουμε σε καινοτομίε που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και ανάκαμψη έτσι Ευρωπαϊ... Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν ένα πιο φιλόδοξο πακέτο για την οικονομία την κυκλική και να μπορέσουμε να δράσουμε ταυτόχρονα για το περιβάλλον κ. Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή κοινωνία καταναλώνει ανανεώσιμους πόρους κατά 50% ταχύτερα από ό,τι μπορεί να τους αντικαταστήσει. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει έξι φορές περισσότερες ύλες και φυσικούς πόρους από ό,τι εξάγει εισάγει επομένως έξι φορές περισσότερες ύλες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί μια κυκλική οικονομία με κανόνα την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Απέναντι στο γραμμικό σύστημα κατανάλωσης, το πακέτο μέτρων της κυκλικής οικονομίας είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η κυκλική οικονομία θα πρέπει να δώσει και οικονομικά ωφέλη. Και αυτό θα το καταφέρει εάν την εφαρμόσουμε μέχρι το 2030. Οπότε θα μειωθούν οι δαπάνε κατά 600 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως τα συνολικά ωφέλη θα φτάσουν το 1,83 εκατομμύρια ευρώ. Θα δημιουργηθούν 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά. Τέλος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030 θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα, την επιστήμη για να προωθηθεί έτσι το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ποντάρουμε στην κυκλική οικονομία μαζί με την ισότητα και ε, την ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται όσο καμιά άλλη περιφέρεια του κόσμου από την εισαγωγή πρώτων υλών. Ε, είναι πόρος λοιπόν και τα απόβλητα θα πρέπει να ποντάρουμε ε, και να ε, επενδύσουμε ε, σε κλάδους που μας επιτρέπουν μέχρι και 70% εξοικονόμηση των πόρων, βιώσιμη ανάπτυξη, ευφυή e e, με 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό είμαι υπέρ δεσμευτικών στόχων ανακύκλωσης, υπέρ της κατάργησης όλων των χιτή και των χιτά και θα πρέπει να γίνει σήμα κατά τεθέν στην Ευρώπη και του Made in Europe. Μια κοινή φορολογική πολιτική που να στηρίζει την κυκλική οικονομία, παραγωγή βιώσιμη να ενισχύεται απέναντι σε εκείνη που δεν είναι βιώσιμη. Επιπλέον, στα φορολογικά συστήματα θα πρέπει να μπει και μια κλίδα ε, επαναχρησιμοποίηση. Ευχαριστώ, κύριος Thank you very much. Ε, Φάναγκαν. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Γι' αυτό η κυκλική οικονομία είναι παραπάνω από νομοθεσία και λόγια για την κυκλική οικονομία. Μια κυκλική οικονομία θα πρέπει να έχει να κάνει με τον τρόπο που ο καθένα ζει και που είναι υποχρεωμένο να ζήσει. Αν θέλουμε να γίνει αυτό, ένα από τα πρώτα πράγματα που ε, πρέπει να κάνει κάποιο είναι να δίνει το παράδειγμα. Μπορούμε να αναρωτηθούμε, δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα, πώς ζούμε, ε, κάνουμε ε, ανακύκλωση, μείωση και τα λοιπά αποβλήτων καθόλου. Κοιτάξτε τι γίνεται με το νερό που πίνουν εδώ οι βουλευτές, είναι σε πλαστικά μπουκάλια. Τι θα γίνει, κοιτάξτε τις μηχανές του καφέ. Εκεί πέρα έχουμε κάψουλες που σχεδόν δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Ε, ε, δεν σας φτάνει να έχετε μια κανάτα καφέ ε, ε, και κουταλάκια. Ε, πάμε Στρασβούργο κάθε μήνα. Αυτό το λέτε μείωση των εκπομπών. Εγώ πηγαίνω σε επιτροπές. Ζητάμε από τον κόσμο να μας παρακολουθεί και βλέπουμε χιλιόμετρα χαρτιά. Έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη mail. Ε, πώς θα δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριο Σέκχαουτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο θα αναρωτιέστε γιατί είμαστε τόσο επικριτικοί, γιατί εδώ πρόκειται για την αξιοπιστία της Κομισιόν. Είχατε υποσχεθεί να, είμαστε, να είσαστε πιο φιλόδοξοι. Τώρα τι γίνεται. Έχουμε ένα σχέδιο δράση, έχουμε μια δήλωση, έχουμε μια στρατηγική, έχουμε οδικό χάρτη, έχουμε πολλά για την κυκλική οικονομία, αλλά αυτό το σχέδιο δράσης κατά τι διαφέρει από τα προηγούμενα. Δεύτερο, για το νομοθετικό πακέτο γιατί χρειάστηκε να αποσυρθεί πριν από 1,5 χρόνο, διότι το μόνο που προσθέσατε από τότε είναι το σχέδιο δράσης. Γιατί χρειάστηκε να αποσυρθεί τότε. Όσο για το περιεχόμενο βλέπουμε χαμηλότερους στόχους, λιγότερους στην νομοθετική πρόταση και ένα σαφές ερώτημα. Πού είναι ο στόχος για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων μας. Αυτό έχει σβηστεί και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ. Μπόγκοβιτς. Βιτσίπα. Ευχαριστώ. Η κυκλική οικονομία είναι η σωστή απόφαση και υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν μέσα στις διορίες που είχε ανακοινώσει. Θα πρέπει να αποτελέσει ένα νέο πρότυπο και όχι απλώς μια σωρία εγγράφων. Πρέπει να βιωθεί, να εφαρμοστεί και κατά την εφαρμογή της πρέπει να βασιστούμε στους ανθρώπους διότι τα άτομα θα αποφασίσουν πόσα τρόφιμα θέλουν να φάνε και πόσα θα πετάξουν και τα άτομα αποφασίζουν τι θα κάνουν με τα απόβλητα. Να στηριχτούμε λοιπόν στους νέους που μπορούν να προωθήσουν αυτού του είδους την οικονομία και που θα είναι εκείνοι που θα ζήσουν τη νέα αυτή οικονομία. Γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω ότι συζητούμε τους στόχους αλλά ιδιαίτερα πρέπει να τους βιώσουμε τους στόχους της κυκλικής οικονομίας. Ο κύριος Σεράος Σάντος. Ευχαριστώ. Ένας από τους στόχους ε, της εφαρμογής ε, αυτής της κυκλικής οικονομίας είναι η διαχείριση των αποβλήτων, ε, των οποίων ο αντίκτυπος στην θάλασσα και όχι μόνο είναι πολύ πολύ σημαντικός. Το πλαστικό και κυρίως το μικροπλαστικό είναι αυτό που δημιουργεί μέγα πρόβλημα για την, την μόλυνση των, οργαν, θαλασσίων οργανισμών. Προκαλούνται ορμονικά προβλήματα που στρεβλώνουν τα ποσοστά ανάπτυξής τους και αναπαραγωγής τους. Ε, είναι υπεύθυνα για την, ε, ε, για την μείωση της αναπαραγωγής πολλών ειδών θαλασσίων θηλαστικών αλλά και ψαριών. Όλα αυτά δεν είναι λύση. Λύση είναι η γρήγορη υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε και τώρα επαναρχόμαστε στον κύριο Κατάινεν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τις συμβουλές σας. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι ο Επίτροπος θα έρθει στις 21 ε, Δεκεμβρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να μελετήσετε τα θέματα αυτά εκτενώς και σε λεπτομέρειες. Πρώτον, τι αλλάζει σε σχέση με το παρόν πρόγραμμα και μάλλον με το προηγούμενο, ε, την προηγούμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προηγούμενη πρόταση νομοθετική για τα απόβλητα ε, βασιζόταν σε ε, κάποιους στόχους που ήταν ευχολόγια. Δεν ήταν νομικά δεσμευτική η στόχη, ας πούμε, για την χωματήρη και καμία πολιτική ομάδα, ούτε οι πράσινοι ε, θα ε, πόνταραν στην αλλαγή που θα ήταν λιγότερο ε, φιλόδοξη από αυτό που προτείνουμε. Ήταν ευκολόγιο, ήταν κάποια ελπίδα που εκφράσαμε ότι κάποιος μπορεί να το κάνει. Τώρα αυτό που προτείνουμε είναι νομικά δεσμευτικό. Και μάλιστα όχι 25% αλλά 10% μέχρι το 2030. Επίσης, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι δεν συζητούμε μόνο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα απόβλητα, αλλά πώς και θα μειώσουμε την παραγωγή αποβλήτων. Αυτό είναι σημαντικό και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θελήσαμε με το πακέτο αυτό και τη δέσμη να έχουμε πιο ρεαλιστικές και πιο φιλόδοξες προτάσεις για να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε την παραγωγή αποβλήτων. Να μειώσουμε τις ποσότητες αποβλήτων και να ε, χρησιμοποιήσουμε και κίνητρα για να ε, χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα απόβλητα που είναι πολύτιμη πρώτη ύλη για τη βιομηχανία. Άρα, ε, χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τον κύριο Ταγιάννη να χρησιμοποιεί τον όρο επαναβιομηχανοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εκβιομηχάνηση της Ευρώπης, γιατί είναι σωστά τα κίνητρα που δίνουμε. Το είπε και άλλος ο κ. Ντέλιτσλα για τους ε, οικονομικούς στόχους και τα κίνητρα. Εάν ε, το καταφέρουμε με το σωστό τρόπο, πραγματικά ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα, τους επιχειρηματίες και την καινοτομία και την βιομηχανία να ε, έχουν ένα άλλο επιχειρηματικό μοντέλο προς την κυκλική οικονομία περισσότερο. Επίσης, αν συγκρίνουμε τους στόχους για την ανακύκλωση με τους στόχους για το χιτά και χιτή, είναι μία ενότητα. Μέχρι το 2030 η ανακύκλωση θα πρέπει να έχει φτάσει στο 65% και είναι νομικά δεσμευτικό, επαναλαμβάνω, και έχουμε και νέους στόχους, δηλαδή μέχρι το 2025 θα πρέπει να κοιτάξουμε αν θα χρειαστεί να αυξηθεί ο στόχος αυτός ε, πάνω από το 65%. Όταν αλλάξαμε και το στόχο για τις χωματερές, για να είναι πιο φιλόδοξος. Ε, αυτό ε, είχαμε υπόψη μας, να υπάρχει μεγαλύτερη ανακύκλωση. Ε, πόσες θα είναι οι θέσεις εργασίας, ό,τι γνωρίζει. Έχουμε υπολογίσει ότι αν δούμε μόνο το στόχο για την ανακύκλωση και για τις χωματερές, είναι περίπου 170.000 νέες θέσεις εργασίας άμεσες. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει το μοντέλο της οικονομίας στο μεταξύ. Αν δείτε τον οικολογικό σχεδιασμό και την αντίστοιχη οδηγία ή τις πρακτικές ή ε, την ε, ε, σήμανση της ενέργειας, χωρίς να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής, με τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή, τι διαπιστώνουμε και τι εκτιμούμε. Ότι μέχρι το έτος 2020 η ενέργεια που θα έχει εξοικονομηθεί θα είναι περίπου η ίδια με την ετήσια ε, πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας της Ιταλίας. Βασικά δηλαδή εξοικονομούνται και χρήματα και αυξάνεται η αγοριστική δύναμη του μέσου καταναλωτή στην Ευρώπη τουλάχιστον κατά 500 ευρώ το χρόνο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να υπολογίσει τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και ακόμα μπορούσαμε και αν προσθέσουμε ε, Ε, αυτό και στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε για τη συζήτηση αυτή. Ένα τελευταίο για τη σπατάλη τροφίμων, γιατί ακούστηκε από πολλούς. Τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί για ε, τους στόχους αυτούς για την βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό το λέει και το νομοθετικό πακέτο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πάρουν εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται για να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων σε κάθε χώρα και να ελέγχουν ε, την ε, διατροφική αλυσίδα για να υπάρξει πρόοδος. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει μια κοινή μεθοδολογία για να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Έτσι ε, θα έχουμε και ενιαία νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Και μάλιστα αυτό θα βοηθήσει προς μια κυκλική οικονομία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να διατίθενται τα τρόφιμα και να μην ε, πετιούνται. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Υπάρχει πολλή χώρο για ρεαλιστική, πραγματική ε, προσέγγιση, μέτριοπαθή, στοχευμένη, ε, με στόχο τα αποτελέσματα, τα απτά και τα συγκεκριμένα. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε νέα μέτρα για να μπορέσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να έχουν εκείνη τη δύναμη να αλλάξουν το μοντέλο το οικονομικό μας. Ευχαριστώ.